Giovanni Lavia, che ne ha facoltà. Ο κύριος Τζοβάνι Λαβία Είμαι υπέρ του συμβιβασμού που επετεύχθη για την πρόταση οδηγίας